αποχές απορρίπτεται 287 και άγκρι 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία διακόπτει ο πρόεδρος άγκρι 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 290 του συναδέλφου Πότς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίες 292 και άγκρι 51 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 293 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη συμβαστική πρόταση 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 299 και άγκρι 55 που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική πρόταση 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 305. Ποιος είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 337 τροπολογία τώρα. Ποιος είναι υπέρ. 337 Πεντητσίνη, Αφρόντε και Εύη, οι συνάδελφοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 338. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 339 και άγκρι 66. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 340. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 341 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 342 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 347 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 348 και άγκρι 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 349 και άγκρι 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 350 και άγκρι 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 351 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 359 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 362 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος κουραστήκατε λέει ο πρόεδρος άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε τώρα στην 372 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 374 υπέρ κατά επαναλαμβάνω λέει ο πρόεδρος επαναλαμβάνω και πάλι υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία τώρα 375 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 376 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 377 και άγκρι 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 378 υπέρ είναι συμβατό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογίες ταυτόσημες 381, 382 και άγκρι 74 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 399 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 400 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 401 και άγκρι 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 402 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία άγκρι 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 405 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 406 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες 408 και άγκρι 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 410 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 411 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 418. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 419. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 421 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 πρέπει να ψηφίσουμε. 422. Ποιος είναι υπέρ του 422. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Α, έλεγχο θέλετε. Ωραία. Για την 423 τροπολογία. Ελέγχουμε. Ψηφίστε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε Διακόπτη Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 37, τροπολογία 37, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 424, καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε το συμβιβασμό 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική πρόταση 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 435 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία, διορθώνει ο συμβαστική πρόταση 32 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 436 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψηφό. Συμβαστική πρόταση 31. κατά αποχές εγκρίνεται. 33 συμβαστική πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 44, τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 92 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 458 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 459 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά αποχές συγγνώμη Η πράσινη και η γκου εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται ας αλέξουμε λέει ο πρόεδρος ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορίας σαφή, ξεκάθαρη πλειοψηφία. Στο συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. 461, 462 και άγκρι 93 τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 464. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 465 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 466 και άγκρι 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 467 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 469 και άγκρι 97 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία ε, άγκρι 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 471 υπέρ. Κατά Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο. Διαφορά. Άγκρι 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 100. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 473 και άγκρια 101 ταυτόσημες υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψήφισατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Προπολογία 474 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 475 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 476 και άγκρη 103 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτονται. Έλεγχος. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει ο Πρόεδρος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 49 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 477 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνετε; 478 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 481 481 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 104 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 482 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβατή 483 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 484 υπέρ. 484 και 493 μαζί λέει ο Πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Άγκρι 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 494 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 495 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 496 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 497 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογίες 498 και άκρη 108 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 499 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 501 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 502 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 503 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 504 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 505 και 506 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 507 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 508 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 509 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 510 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 511 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 512 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 513 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 514 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 35 υπέρ. Κατά αποχές με ναι, εγκρίνεται. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία της συμβαστικής πρόταση 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 563 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 562 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 564 λέει ο πρόεδρος αλλά διακόπτη θα πρέπει να ψηφίσουμε την 561 δεύτερο τμήμα της τροπολογίας της συναδέλφου Λίζε. Συμβαθεί, δηλαδή με 563 και 562 τροπολογίες. Η γραμματεία λέει ότι πρέπει να την ψηφίσουμε. 561 λοιπόν δεύτερο τμήμα τη τροπολογία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 564 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 565 και άγκρα 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 566 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Έχουμε έναν σοσιαλιστή παραπάνω, λέει ο Πρόεδρος. Ψήφισατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την 567 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία όχι, λέει πρόεδρος, πάμε κατευθείαν στην συμβαστική πρόταση 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 591 συναδέλφου Λίζε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 592 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μάλλον θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λέει ο πρώτος έλεγχο. Ψήφισατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 593 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 συμβατή με την 593 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την 598 του Σανδέλφου Πότς. 598 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 597 καθώς και την <clears throat> Άγκρι 118, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η Άγκρι 118, <clears throat> δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 599 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 που είναι τα συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 600 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 601 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 602 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 603 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 65 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 604 <clears throat> υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.15 υπέρ κατά αποχές απορρίζεται 616 και 616 και 122 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίζεται 6-17 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, <clears throat> απερίφθη. 6-19 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Ισοψηφία. Απορρίψετε. 618 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 620 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται 621 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τσεκ, βεβαίω. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 623 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 624 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 627 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 123 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 641 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.42 και άγκρι 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 6.44 και άγκρι 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 6.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.43 έλεγχος υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, <clears throat> εγκρίθηκε. 6,40, 130 άγκρι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 658 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 661 υπέρ 661 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 662 είναι σημαντική, υπέρ κατά αποχές Απολύτωται. 663 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, Απολύτωται. 664 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 665 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 666 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας απερίφθη. 667 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας απερίφθηκε 668 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 669 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 670 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 671 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 672 και 673 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνονται 674 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 675 υπέρ 1 κατά αποχές εγκρίνονται. 676 και 677 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 678 679 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, ισοψηφία απορρίπτονται. Τώρα, 680 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 681 υπέρ κατά αποχέ το ΙΣΙΑ δεν ψηφίζει έλεγχος 681 Χρειάζομαι την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Συζητάτε όλοι, όλες. <clears throat> Πέρας. Εγκρίνεται. 682. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 683 και την 134 άγκρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 684 και άγκρη 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 686 και άγκρη 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 687 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 688 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 689 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. <clears throat> εβδομήντα 72 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. <clears throat> 692 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 693 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Καλά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Εβδομήντα πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 694 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πάμε στην τροπολογία 100 δεύτερο τμήμα Κάντεμπαχ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 709 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασκή 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.30 3 που είναι, είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 734 και 737 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 741 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 740 και 742 και 7.43 επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 7.44 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 762 δεύτερο τμήμα. 72, συγγνώμη. Κατά αποχές εγκρίνεται. 775 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος είναι 775. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 784. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 787 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, απορρίπτεται. 788 υπέρ αυτά αποχές έλεγχος. Εφτά, οχτώ, οχτώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εφτά 7, εφτά και 7, 98 είναι εκεί υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 7-9 <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 800 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 801 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 802 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 803 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 804 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 821 και 829 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. απορρίπτεται. Συμβασική 17 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 154 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Οκτώ Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 155. Υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 8.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 867 υπέρ τα αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται Άγκρι 156 και 868 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται έλεγχος βεβαίως Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκαν 869 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 870 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 Άγκρι 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται 871 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 872 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 873 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 874 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 875 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται 876 υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 159 υπέρ κατά αποχές Πού είναι οι σοσιαλιστέ. Υπέρ ή κατά. Υπέρ. Εντάξει, εγκρίνεται. 8.93. Εκπίπτει. Πάμε στην 8.89. 8.89. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8.90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8.91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.92 υπέρ κατά έλεγχος Όλοι ψηφίσατε. Πέρασε. Απόλυτα. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 894 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 895 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 105 σε δύο δόσεις, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 899 και 162 που είναι άγκρι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 900 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 901 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 902 υπέρ 902 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 904 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι ψηφίζουμε τώρα. 905 καθώς και άγρια 166. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 906 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 907 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 908 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 909 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 910 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 911 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 912 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απολύτωται. απότε. μια δεκαέξι, ψηφίσουμε από κοινού. <clears throat> ναι, μαζί τέσσερις υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 918 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκα... 9, και 167 άγκρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 9-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 9-21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9-22 υπέρ κατά έρχος Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 9.23. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 924 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωση 925 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωση 926 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωση 927 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωση 928 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 929 <clears throat> υπέρ κατά απόχες ελέγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας απορρίπτεται με ισοψηφία. 9.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 933 και αγκρί 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 934 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίφθηκε. 935 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9.36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε 9.37 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Εγκρίνεται. 9.38 υπέρ. Κατά αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται αλλά στο ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 9.39. Υπέρ. Κατά. αποχή, Εγκρίνεται. 9.40. Υπέρ. Κατά. αποχή, έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. περά, Απορρίπτεται. Votiamo il 900. 941. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 942 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 943 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. όλοι, πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 944 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 945 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 946 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατό εφτά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατό οχτώ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Εκατό εννέα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατό δέκα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγκριένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 που είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 125 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άγκρι 5 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά απόχέ. απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 130 και άγκρι 6 ταυτόσημε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 131 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ο πρόεδρος έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρα στις πληροφορίες απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, 154 κατά πίπτη, 156 ψηφίζουμε, 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 159 όχι, Άγκρι 10. Άγκρι 10. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος λέει ο πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 164 και άγκρι 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 12 καταπίπτει, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος καταπίπτει η άκρη 12 ποιοι κάνουν 168 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στην 171 γιάρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε την άκρη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άγκρη 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές τα ελέγξουμε λέει ο ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ψήφισατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 και άγκρι 15 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τον 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος λέει ο πρόεδρος ψήφισατε όλοι πέρας Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Συγγνώμη, ο Λεοπρόδος διορθώνει. 185 πρέπει να ψηφίσουμε. 83-84 καταπίπτουν. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 19 υπέρ κατά, α, κατά αποχές θα ελέγξουμε λέει πρόεδρος ψήφισατε όλοι πέρας απορρίπτεται Ψηφίζουμε την 189 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκρή 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 καταπίπτει θα δούμε στη τελευταία σελίδα 195 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ψήφισατε όλοι πέρας απορρίπτεται 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος λέει πρόεδρος. Ψήφισατε όλοι. Περάς. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 31-31. Ψηφίζουμε τώρα την Άγκρη 22 υπέρ. Άγκρη 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198 και Άγκρη 23 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 199 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 201 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ο λόγος είναι συγγετρία. Ναι. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους συναδέλφους για την υπομονή. Ήταν μακροσκελής αυτή η ψηφορία. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Ήταν δύσκολο να προεδρεύσει κανείς όταν έχουμε τόσες τροπολογίες να ψηφίσουμε. Να ψηφίσω λοιπόν τους συναδέλφους, αλλά κυρίως τους σκιώδεις από τις πολιτικές ομάδες γιατί όπως είδατε είχαμε πολλές συμβαστικές τροπολογίες που απέτησαν πολλές συνεδριάσεις για άρθρα αρκετά περίπλοκα κάποιες φορές. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους για την ατμόσφαιρα υπό την οποία κάναμε αυτή τη δουλειά και την πολύ καλή συνεργασία. Ομολογώ σήμερα αυτό που υποβλήθηκε είναι μια ομαδική δουλειά που έγινε και θα ήθελα να το τονίσω. Σήμερα δεν θα ήθελα να σας ζητήσω άμεσα εντολή διαπραγματεύσεων για αυτό το κείμενο, επειδή θα επιθυμούσα η έκθεση αυτή να περάσει στην Ολομέλεια, θεωρώντας ότι για ένα κείμενο τόσο σημαντικό, με τόσα διακυβεύματα δημόσιας υγείας, μου φάνηκε σημαντικό να μπορούν να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι και όχι μόνο τα μέλη της Επιτροπής μας αυτής. Οπότε θα σεβαστώ απολύτως το πνεύμα της νομοθετικής διαδικασίας και το ρόλο του Κοινοβουλίου και δεν θα υποχωρήσω ενώπιον της δημόσιας συζήτηση. Είναι νομίζω σημαντικό να μπορέσουμε να περάσουμε την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια ή του Μάρτη ή του Απρίλη. Εν τω μεταξύ, έχω ακόμα άλλο ένα μήνυμα να σας στείλω, δηλαδή ότι δουλέψαμε πολύ για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα και βεβαίως γνωρίζω ότι όπως κάθε συμβιβασμός αυτή η έκθεση ήταν αντικείμενο πολλών συμβιβασμών που βεβαίως δεν ικανοποιούν απολύτως τους πάντες. Αυτό είναι προφανές. Αποτελεί τον καρπό των προσδοκίων του καθενός. Και εκ μέρους μου χαίρομαι, ξαναλέω, επειδή αυτή η δουλειά ήταν περίπλοκη, την οποία όμως κάναμε από κοινού και θα επιθυμούσα να υιοθετηθεί στην Ολομέλεια και να μπορέσουμε τότε να έχουμε ως τελικό αποτελέσμα ένα ισχυρό κείμενο, συνεπές κείμενο και ευανάγνωστο κείμενο. Γιατί, όπως έλεγα, τα διακυβεύματα που αφορούν δημόσια υγεία είναι πολύ σημαντικά. Αν πάμε λοιπόν στην Ολομέλεια, το μήνυμα που έχω να σας στείλω είναι ότι όλοι μας θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα, ώστε να μην επαναυποβάλουμε, να μην επανακαταθέσουμε τις τροπολογίες οι οποίες απορρίφθηκαν σήμερα, γιατί πραγματικά διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε ένα κείμενο που θα χάσει σε συνέπεια και σε ισορροπία. Θα ξαναζητήσουμε, το ξέρω και χαίρομαι. Όμως ε, θα ήθελα να μην ε, διακινδυνεύσουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει ε, με τόσο κόπο και πάλι ευχαριστώ όλους τους κοιόδης όλων των πολιτικών ομάδων, αλλά ευχαριστώ και όλους τους συμβούλους μας ε, που μας ε, βοήθησαν. Αυτά είχα να πω. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, εάν συμφωνούν και οι συνάδελφοι, να στείλουμε αυτό το κείμενο προς ψηφοφορία, στην, ε, προς ψήφιση μάλλον, στην Ολομέλεια. Και σας ευχαριστώ όλους. We have now... Εντάξει. Έχουμε τώρα την τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα ηλεκτρονικά, οπότε άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην εισηγητρία. tanto la presentazione in 10 minuti non facciamo il eh. ah, ah, ah, Now we go to the next point in our agenda. It is... Uh, Επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Ε, τι. Άψη φορία είναι πάλι. Λοιπόν, για, η επόμενη ψηφοφορία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο κύριος Τανασέσκου είναι εισηγητής. Emendamento 24. 24. Με προφορική τροποποίηση έχετε αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση. Όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 με προφορική τροποποίηση των πρασίνων υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 με προφορική τροποποίηση από το ΕΛΚ. Αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίσουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 και 28 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 άγκρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 με προφορική τροποποίηση από το ΕΛΚ. Υπάρχουν αντίρρησεις. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 με προφορικές τροποποίησεις από το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές. Αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε 33 με τροποποίησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία άγκρι 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρια 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 37 και άγρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 40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 κατά από χες εγκρίνεται 14 υπέρ κατά από χες εγκρίνεται 51 υπέρ κατά από χες απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγκρί 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε σε λογική σκέψη. Αγκρί 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές <clears throat> απορρίπτεται τροπολογία 1 και άγκρη 3 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 με προφορική τροποποίηση υπάρχουν αντιρρήσεις όχι ψηφίζουμε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 σε δύο τμήματα. <clears throat> Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέας απορρίπτεται. Τροπολογία 22 <clears throat> με χωριστή ψηφοφορία και πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά από χες απορρίπτεται. Τροπολογία 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, χές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ο εισηγητής με το λόγο αν θέλει, όχι, τελική ψηφοφορία όπως έχει τροποποιηθεί η πρόταση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 54 εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται. όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε φτάσει στο τέλος των ψηφοφοριών. Έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μέσα διάταξη. Ο κύριος Μπερτολίνη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να μας κάνει την εισήγηση. Δεν θα έχουμε χρόνο ε, να συζητήσουμε μετά, αλλά είναι σημαντικό να γίνει αυτή η πρώτη παρουσίαση και μετά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Dear colleagues, we start immediately. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε κατευθείαν με το επόμενο σημείο. Το λόγο έχει ο κύριος Μπερτολίνη από τον ΠΟΗ για να μας κάνει παρουσίαση στο διαθέσιμο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Τη διαφάνειες παρακαλώ θα ήθελα. Λοιπόν, εν συντομία θα μιλήσω ε, για αυτή τη ε, νέα διεθνή κρίση για τη δημόσια υγεία όπως έχει προκυρηθεί από τον ΠΟΗ από την 1η Φεβρουαρίου που αφορά τον ιό ΖΙΚΑ. Ο ιός ζήκα λοιπόν είναι μια οικία ασθένεια που ε, μεταδίδεται μέσω ενός ε, είδους ε, κουνουπιού. Είναι σημαντικό να πούμε ότι μόνο ένα στους τέσσερις που πλήττονται από τον ιό έχουν συμπτώματα. Και μάλιστα τα συμπτώματα αυτά είναι πολύ ήπια, πυρετός, εξάνθημα, μυϊκή πόνη, επιφυγίτιδα. Δεν υπάρχει όμως θεραπεία ή εμβόλιο. Γιατί όμως πληγρήθηκε η κατάσταση της επίγουσας ε, κρίσης είναι ε, οι περιπτώσεις ε, μικροκεφαλίασης που είναι δηλαδή ότι ένα παιδί που γεννιέται με πολύ μικρό κεφάλι λόγω ελλειπούς ανάπτυξης του εγκεφάλου. Και υπάρχει και ένα άλλο σύμπτωμα που το οποίο αφορά τους ε, ενήλικες, τους νέους ενήλικες, ε, που προκαλεί αδυναμία του ε, ανοσοποιητικού και παράλυση. Η πλειονότητα όσων πλήττονται από τον ιό ουσιαστικά τους τσιβάει το κουνούπι και έχουμε πολύ μικρά περιορισμένα στοιχεία για άλλες διόδους μετάδοσης του ιού. Νομίζω υπάρχουν τρεις περιπτώσεις ε, στη βιβλιογραφία που καταδεικνύουν σεξουαλική μετάδοση ε, από άντρα σε γυναίκα. Ένας άντρας δηλαδή που έχει πληγεί από τον ιό ε, μέσω σεξουαλικής επαφής μεταδίδει τον ιό σε γυναίκα. Και ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω αίματος. Όταν γίνεται μετάγγιση αίματος μπορεί να μεταδοθεί και ο ιός. Ο κύριος μηχανισμός τώρα και τρόπος προστασίας. Είπα ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε υπάρχει εμβόλιο. Οι ταξιδιώτες ε, μπορούν να προστατευθούν με τους συνήθεις τρόπους ε, που χρησιμοποιούν για να αποφύγουν τα τσιμήματα από κουνούπια, όπως είναι τα έντομα τα ανοιχτόχρωμα ρούχα, ε, εμπόδια όπως είναι οι πόρτες και τα παράθυρα να μένουν οι κουνουπιέρες και ε, να αδειάζουμε ή να καλύπτουμε ε, μέρη όπου συνήθως βαλτώνουν νερά και εκεί μπορούν να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν τα κουνούπια. Τώρα, ε, πρώτα απ' όλα σε μαϊμούδες το είχαμε εντοπίσει τον ιό αυτό στην Ουγγάντα το 1947 και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αναπτύχθηκε. Γιατί στην αρχή πήγε στη Δυτική Αφρική, μετά μεταδόθηκε στην Ήπειρο της Ασίας μετά πάλι προς την Ινδονησία, πιο ανατολικά και άλλες νήσους προς τα εκεί, μετά στο Γκουάμ και σε νησιά του Ειρηνικού, το 2007 έγινε αυτό, ε, στην Γαλλική Πολυνησία το 2013, μετά ε, στην ίσο του Πάσχα, στη Χιλή και μετά στη Λατινική Αμερική. Και τώρα έχετε μια επισκόπηση της γενικής κατάστασης, οι χώρες δηλαδή όπου ε, απαντά ο Εδώ έχετε τον κατάλογο των χωρών που έχουν πληγεί, περίπου 34 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού. Τώρα, βλέπετε και την ανάπτυξη σε χρονικό πλαίσιο ε, που μας δημιουργεί και αυτή την ανησυχία. Γιατί εντοπίσαμε τις τα πρώτα κρούσματα του 2015, το Μάιο, επιβεβαιώθηκαν λίγο αργότερα, πάλι το Μάιο. Μετά είχαμε ε, στην Παΐα της Βραζιλίας τον Αύγουστο του συνδρόμου Γκυγιάν Βαρέ. Μετά και η Κολομβία ανέφερε κρούσματα. Ε, στις 30 Οκτωβρίου η Βραζιλία ε, δήλωσε ότι υπάρχει ασυνήθιστη αύξηση της της στη, λόγω του ιού Ζήκα. Και μετά στις 30 Ιανουαρίου 26 χώρε έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν ευεβεβαιωμένες ε, υποθέσεις και έτσι 1η Φεβρουαρίου ε, κρίνουμε πλέον ότι πρόκειται για μια ε, κρίση παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Έχουμε περίπου 4.000, πάνω από 4.000 μάλλον, περιπτώσεις μικροεξεφαλίας στην Βραζιλία και περίπου 1,5 ε, εκατομμύριο ε, περιπτώσεις κρουσμάτων από τον ιό Ζήκα. Αλλά είναι πολύ ήπια τα συμπτώματα. Παναλαμβάνω, πολλές φορές ε, δεν ξέρουν καν οι ασθενείς ότι υπάρχουν. Μετά, κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, στις 30 Ιανουαρίου ο Υπουργός της Βραζιλίας ανέφερε 4.783 υποθέσει υποθέσεις, ακόμα και 76 θανάτους. Όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι από τις 1.100 υποθέσεις που έχουμε αναλύσει σε βάθος, σε 1.100 κρούσματα, γιατί πρέπει να αναλύσουμε όχι μόνο την περίμετρο της κεφαλής, αλλά και με ακτινογραφίες και άλλες ενδείξεις ε, των συμπτωμάτων που συνδέονται με την κεφαλίαση. Μόνο 404 ε, υποθέσεις κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί. Τα υπόλοιπα ε, έχουν απορριφθεί. Και τα υπόλοιπα 3.670 κρούσματα ακόμα διερευνώνται. Επομένω, είναι πιθανό μόνο το 1 τέταρτο αυτών των 4.000 πλέον ε, ε, κρούσματων να είναι όντω μικροκεφαλίαση. Και σε αυτή την περίπτωση και πάλι είναι πολύ αυξημένο ο αριθμό ε, για τη Βραζιλία. Γιατί συνήθω είναι 200 περιπτώσει τον χρόνο στη Βραζιλία. Έχουμε λοιπόν πενταπλάσιο ή δεκαπλάσιο αριθμό κρουσμάτων. Σίγουρα υπάρχει λοιπόν ε, ένα επιδημικός πυρήνας. Λοιπόν, σε 17 κρούσματα εντοπίστηκε ότι όντως πρόκειται για τον ιό Ζήκα, από τα 387 δηλαδή, και να υπογραμμίσω ότι στην Γαλλική Πολυνησία που είχε μια επιδημία από το 13 στο 14 υπήρξαν βρέφη τα οποία γεννήθηκαν με γενετικές ανομαλίες. Δεν είναι κάτι καινούριο λοιπόν. Τώρα έχουμε αυτή την επιδημία και στην Βραζιλία. Δεν είναι όμως η, πρώτη περίπτωση που έχουμε ε, κρούσματα μικροκεφαλίασης. Όμως το σημαντικό είναι σε μια περίπτωση στη Σλοβενία που έχει παρατηρηθεί ε, Μία γυναίκα λοιπόν που είχε ε, πληγεί από τον ιό Ζήκα στη 13η εβδομάδα γεμοσύνης της όταν εργαζόταν στην Βραζιλία. Ε, επέστρεψε στη χώρα της λοιπόν, στις 28 εβδομάδες ε, εντοπίστηκε η μικροκεφαλία της στο, στο έμβριο και προχώρησε σε τερματισμό της κοίησης και εκ των υστέρων ε, όντως ε, διαγνώστηκε ότι υπήρχε μικροκεφαλίαση, ότι είχε πληγεί από τον Ζήκα. Είναι λοιπόν βέβαια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά είναι σημαντική. Τώρα, 1η Φεβρουαρίου, όπω είπα, είπαμε ότι υπάρχει ε, διεθνής κρίση και συνδέεται με την υποψία σύνδεση μεταξύ ΖΙΚΑ και μικροκεφαλίασης. Είναι έκτακτη κατάσταση και απαιτείται μια διεθνή συντονισμένη δράση. Παρότι υπό τους διεθνείς κανονισμούς ο ΠΟΗ μπορεί να ε, αναφέρει συγκεκριμένες ε, ε, περιορισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, αυτό ισχύει μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις γυναικών να μην ταξιδεύουν αλλού κτλ. Έχω συνοψίσει κάποια από τα κύρια ζητήματα. Έχουμε πολλά νέα στοιχεία, υπάρχει αβεβαιότητα για κάποια στοιχεία. Πρέπει να αναπτύξουμε εργαστηριακούς ελέγχους που ακόμα ε, δεν είναι ε, πλήρως ε, διαθέσιμοι. Υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά την κλινική εποπτεία όπου υπάρχει υποψία μικροκεφαλίας Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τέτοιες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τον τερματισμό και και αν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ε, ο έλεγχος ε, των φορέων του ιού, τα μέτρα δηλαδή που θα υιοθετηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και σε ό,τι φορά την ε, απολύμανση των αεροσκαφών που έρχονται από αυτές τις ε, μολυσμένες χώρες. Ο κίνδυνος ε, των, ε, των ταξιδιωτών από αυτές τις χώρες προς την Ευρώπη σίγουρα αυξάνεται, όμως αυτό το, το είδος κουνουπιού, το AIDS, δεν το βλέπουμε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης ε, του ιού ε, στην Ευρώπη. Αν και την άνοιξη και το καλοκαίρι ε, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η μετάδοση του ιού στην Ευρώπη γιατί είναι καλύτερο το κλίμα. Τώρα, το a που είναι ο, η, μορφή του κουνούπιου, ο τύπος του κουνούπιου αυτού, βλέπετε ότι παρέχεται στην Ευρώπη μόνο σε αυτή την περιοχή στο κόκκινο, το ανατολικό τμήμα της ε, ε, Μαύρης Θάλασσας. Όμως το Αλμπουπίκτους, που είναι ένα άλλο κουνούπι, το λεγόμενο κουνούπι Τίγρης, ε, μεταδίδει και τον ιό Τσικαγκούια. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε αυτό τον ιό που υπήρχε μια επιδημία στη Ραβένα της Ιταλίας του 2007, είχαμε περίπου 300 τέτοιες περιπτώσεις Επομένω, ε, υπάρχει ευρεία παρουσία αυτού του κουνουπιού ε, στην Ευρώπη, στην Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Νότια Γαλλία, Ισπανία και κάποιες μεμονωμένες ε, ομάδες κουνουπιών βρίσκονται ακόμα και στην Τσεχία, στις Κατοχώρες χώρες και Επομένως, αν κάποιος με τον ιό έρθει με την ασθένεια έρθει στην Ευρώπη, ε, τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, πάρει το κουνούπι τον ιό και τσιμπήσει κάποιον άλλον, τότε και πάλι μπορεί να υπάρξει η μετάδοση του ιού και αλλού. Όμως, αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σίγουρα θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να ε, ελέγξουμε και να περιορίσουμε την μετάδοση. Και όταν ξεκίνησε αυτή το ε, αυτό αυτή η επιδημία ε, στην Ιταλία, υπήρξε πολύ έντονη ανταπόκριση ε, και ταχύτατη ανταπόκριση του συστήματος δημόσιας υγείας και μέσα σε μερικές μέρες μόνο είδαμε ότι μόλις 200 περίπου τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν. Επομένως, ο δημόσιος κλάδος ανταποκρίθηκε και περιόρισε στο έπακρον την εξάπλωση του Πρώτον, ο έλεγχος λοιπόν ε, της μετάδοσης των φορέων. Είναι σημαντικό αυτό και για το παρόν και το μέλλον. Επικοινωνία, η ενημέρωση των ε, ταξιδιωτών. Να, μην, να αποφεύγουμε όσο γίνεται την επαφή με αυτά τα κουνούπια. Να ενισχύσουμε την, ε, τον εργαστηριακό εντοπισμό και ανείχνευση του ΖΙΚΑ, να ενισχύσουμε την έρευνα και στη διάγνωση και στον εμβολιασμό, ιδίω εάν συνδυαστεί και με την εγκυμοσύνη, ε, όπως και με την Ιλαρά ισχύει ναι. Η Ερυθρά. Υπάρχει ένα ζήτημα της απολύμανσης ε, των αεροσκαφών, ο έχει σαφείς συστάσεις ως προς αυτό το ζήτημα. Ξέρω ότι στην Ιταλία ισχύουν, δεν ξέρω αν ισχύουν κι αλλού. Και ενημέρωση του κοινού. Το Ευρωπαϊκό Τμήμα του ΠΟΗ ε, στηρίζει τις ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε διαθεσίσεις για όλα αυτά τα ζητήματα και υπάρχει και ένας ε, πλήρως ενημερωμένος ιστότοπος Ε, εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ενημερωτικό σημείωμα που επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα. Μπορείτε λοιπόν να πάτε εδώ και να, εκεί και να δείτε τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Ευχαριστώ. I think that we to Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον κύριο Μπερτολίνη για την παρουσίαση αυτή στο τέλος της συνεδριασής μα. Λυπάμαι γιατί καθυστέρησε πολύ η ψηφοφορία και δεν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τον χρόνο ούτε τον χώρο και επομένως πρέπει να κλείσουμε τώρα τη συνεδρίασή μας θα ξεκινήσουμε και πάλι αύριο το πρωί και θα επανέλθουμε το μέλλον, στο μέλλον σε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.